So, good morning, colleagues. I opened the, the... Ευχαριστώ πολύ. Ε, ξεκινάμε με την συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ, το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε μία έκθεση με ένα πολύ μεγάλο τίτλο. Η, η συγγήτρια είναι η κυρία Φαγιόν και θα παρουσιαστεί η έκθεση αυτή όπου μιλάμε για έλεγχο προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενα στη μονομερή αναγνώριση από Κροατία και Κύπρο ε, εγγράφων ισοδυνάμων με τις εθνικές ε, τους θεωρήσεις με σκοπό τη διέλευση από την επικράτειά τους ή όταν υπάρχει προθεσμία διαμονής στην επικράτειά τους, η οποία δεν επερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Φαγιόν, ε, πρωτίστως και μετά στους Σκιώδης και στην Επιτροπή. Η κυρία Φαγιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σλοβενικά γιατί το θέμα είναι αρκετά δύσκολο και θα μιλήσω σλοβενικά για να γίνω καλύτερα κατανοητή. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική αυτή πρόταση και την ε, καλή συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις. Η έκθεση αυτή σχετίζεται με την εφαρμογή του μέσου ε, ελέγχου εξωτερικών συνόρων της Κροατίας και της ε, Κύπρου όταν μπήκε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις συνθήκες έπρεπε να εφαρμόσει την πρώτη φάση της Συμφωνίας Σέγγεν. Ε, συνεπώς, η Κροατία, όπως και οι άλλες χώρες προγενέστερα, πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει τον κανονισμό 3 μάλλον 5-3-9 με συγχωρείτε και θα πρέπει να υπάρχει και ένας αρνητικός κατάλογος. Και αυτή η υποχρέωση ισχύει για χώρες όπως επί παραδείγματι το Μαρόκο. Όταν ε, υπάρχει θεώρηση από μία χώρα εντός ε, Σέγγεν, τότε τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να κινηθούν προς την επικράτεια των άλλων κρατών μελών. Γι' αυτό χρειάζεται ένα καθεστώς ε, θεωρήσεων που να αναφέρεται στις χώρες εκτός Σέγγεν και τις θεωρήσεις τους και γενικότερα τις χώρες ε, για τις οποίες ε, δεν ισχύει η Συμφωνία Σέγγεν. Μονομερός λοιπόν μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένες θεωρήσεις που αφορούν την μακροχρόνια ε, διαμονή σε κράτη-μέλη εντός Σέγγεν. Αυτό αφορούσε το Κονγκό, Έφνης, καθώς και τις μακροχρόνιες θεωρήσεις, δηλαδή για μακροχρόνια διαμονή και άλλες άδειες διαμονής που εκδίδουν κράτη-μέλη εκτός, εκτός χώρου Σέγγεν. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο ίσχυε με έναν πολίτη Μολδαβό που η θεώρησή του έγινε αποδεκτή από τη Ρουμανία για στη Ρουμανία, στη διαμονή του στη Ρουμανία. Ο κανονισμός 539 κάθετος 01 αφορά τη μονομερή αναγνώριση των θεωρήσεων που εκδίδονται από κράτη όπου δεν ισχύουν οι κανόνες Σέγγεν, τουλάχιστον όχι πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι Ο κανονισμός 810 κάθετος 2009 δεν ισχύει ως προς τους ε, του, περιορισμούς τους. Ε, υπάρχουν όμως θεωρήσεις που έχουν περιορισμένη επικράτεια, ε, περιορισμένη συγγνώμη, ισχύ στην επικράτεια, όπως έφνη στο κοσυφοπέδιο. Αλλού υπάρχει ευχέρεια διακίνησης ε, εκτός από εκείνους που δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τέτοιες θεωρήσεις περιορισμένες διάρκειας που να αποκλείονται από το μονομερές καθεστώς, διότι έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια του χώρου Σέγγεν. Η διεύνηση αυτού του καθεστώτος δεν σημαίνει επιπρόσθετες υποχρεώσεις στην Κροατία και την Κύπρο. Και αυτή η νομική πράξη δεν αποτελεί παρέκκληση από την Συμφωνία προσχώρησης. Πρόκειται για ένα μη δεσμευτικό καθεστώς και η Κροατία μπορεί να αποφασίσει να χορηγεί θεωρήσεις όπως και πριν από τη Συμφωνία Προσχώρησης και αν η Κροατία και η Κύπρος ε, εφαρμόσουν ένα αμοιβαίως αναγνωριζόμενο καθεστώς, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις θεωρήσεις των άλλων κρατών μελών. έτσι ώστε να ισχύουν σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα αναπτυχθεί περαιτέρω όταν οι χώρες αυτές προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν και υπάρχει υποχρέωση, υπάρχουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς Σέγγεν. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τους εμπειρογνώμονες, τη, γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων, συνέταξα αυτή την έκθεση για να φτάσουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο να αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η τροπολογία υπαριθμών 4 απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει ένα νομικό χάσμα που μπορεί να ανακύψει εξαιτίας ε, της μη αναγνώρισης του κοσυφοπεδίου από την Κύπρο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Εάν η Κύπρος εφαρμόσει τους κανονισμούς αυτούς θα πρέπει να αναγνωρίσει την περιορισμένη, τις θεωρήσεις ε, περιορισμένης ισχύω για τους κατοίκους ε, ε, του Κωσυφοπεδίου, αν και δεν αναγνωρίζει το Κωσυφοπέδιο ως κράτος. Τώρα, ως προς την εφαρμογή των κανόνων Σέγγεν, η ισχύ αυτών των εγγράφων για την ισχύ αυτών των εγγράφων θα υπήρχε ένα νομικό κενό. Άρα αυτή η έκθεση είναι έτοιμη για συζήτηση μετά από διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και αναμένω στη συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επί του θέματος. Ευχαριστούμε την κυρία Φαγιόν. Δεν βλέπω συναδέλφους που να ζητάν το λόγο. Οι σκιώδεις είναι παρόντες από ό,τι βλέπω, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής αν θα ήθελα να μας πει μερικά λόγια. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της με τέσσερις τροπολογίες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι πρώτες δύο διευκρινίζουν το κείμενο της ε, Κομισιόν και χαίρομαι ιδιαίτερα που μας εξήγησε τους λόγους ε, της ε, τροπολογίας 4, την, ε, το υπόβαθρο της τροπολογίας 4, διότι είναι περίπλοκο κείμενο αυτό, αλλά η τροπολογία αυτή είναι, ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πνεύμα της Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 3, έχουμε μία ερώτηση προς διευκρίνηση, διότι εδώ προτείνεται να, να γίνει υπό την επιφύλαξη ενδεχομένων μεταβατικών διατάξεων ε, που έχουν εκδοθεί πριν από την ΟΣΑΝΕ ημερομηνία. Ε, τώρα, σε, ίσως όχι σήμερα, αλλά σε κάποια τεχνική σφίσεω συνεδρίαση θα θέλαμε να ξέρουμε ακριβώς ε, τι προβλέπει εδώ η τροπολογία για να μπορέσουμε να απαντήσουμε κι εμείς και να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, αλλά γενικά πιστεύω ότι η, το πνεύμα της ε, της, της εκθέσεως ευθυγραμμίστε με το δικό μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φαγιόν, ε, προτείνω, επειδή έχουμε τεχνική συνεδρίαση και με τους ε, ε, σκιώδεις εισηγητές να το συζητήσουμε σε τεχνικό επίπεδο αλλά μου επιτρέπετε στο χρόνο αυτό να μπορέσω και εγώ να το ξανασκεφτώ ώσπου να ξανασυναντηθούμε σε εσωτερική τεχνική συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Φαγιόν. Και προχωρούμε στο δεύτερο θέμα. Παρόλο που ε, είναι πρόωρη η συζήτηση, 15 λεπτά έχουμε κερδίσει, αλλά δεν πειράζει, ας προχωρήσουμε στο 15 πρόταση για την ανάπτυξη του συστήματος e-call σε οχήματα. Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος βασίζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ο κύριος Φως θα παρουσιάσει το σχέδιο νομοδότησης. Θα μας ενημερώσει για τις ψηφοφορίες στην Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι οι συντονιστέ ζήτησαν διαδικασία υπό τον ε, ε, κανόνα 50 υπό το άρθρο 50 και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Φως. Ευχαριστώ. Εδώ σήμερα μας απασχολεί το λεγόμενο θέμα των e-call που με την υποστήριξη διαφόρων νομικών πράξεων θα πρέπει επιτέλους να επιτύχουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, δηλαδή μια αυτόματη επίγουσα κλίση σε συγκεκριμένους αριθμούς που υποτίθεται θα λειτουργήσει από το 2015. Γενικά πιστεύω ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να το ε, δεχθούμε, να το υποστηρίξουμε, ότι μπορεί να σώσει ζωές. Βεβαίως ε, προκύπτουν ορισμένα ζητήματα προστασίας δεδομένων και με την γνωμοδότηση αυτή προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς δεν ήταν σαφές και στην δεν ήταν. Εάν αυτό το σύστημα ή κολσά αναφέρεται μόνο σε επίγουσες κλήσεις και θα περιοριστεί μόνο σε αυτές ή αν επιπροσθέτως... Ε, τα, θα χρησιμοποιήσουμε ε, τα e-calls ε, και με στοιχεία προσωπικά ή εμπορικής φύσεως ε, συναλλακτικής φύσεως. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των επιγουσών κλήσεων και των άλλων χρήσεων του e-call. εγώ πιστεύω πριν αποφασίσουμε για δύο συστήματα, να αποφασίσουμε επί της ουσίας της προστασίας δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα είναι ενυπνώσει, ας πούμε, ανενεργό, μέχρι ότου χρειαστεί να δραστηριοποιηθεί μέσω μιας κλήσης. Το σύστημα αυτό δεν θα αποθηκεύει, ούτε θα μεταφέρει ε, δεδομένα, θα μεταβιβάζει δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά την ανείχνευση, το tracking, σε αυτές τις επίγουσες κλήσεις δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να γίνει μια παρακολούθηση, αλλά σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης των ελαχίστων απαραίτητων στοιχείων. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν το σύστημα αυτό να, το, να μπορεί να το κλείσει ο καθένας, ο χρήστης, εάν δεν το εμπιστεύεται. Πρέπει όμως να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση όταν πρόκειται για ιδιωτικής φύσεως ή ε, χρήσης ή άλλης μορφής χρήσης ε, του e-call. Εδώ νομίζω ότι ο νομοθέτης ε, ε, πρέπει να προβλέψει και τα δύο συστήματα παρόλο που αυτή είναι μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσέγγιση. Τα δύο συστήματα θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα τεχνητά τεχνικά και η χρήση του ενός συστήματος δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη χρήση ή να περιορίζει τη χρήση του άλλου συστήματος. Η εισηγήτρια στο ΙΝΚΟ θέλει να περιορίσει τη χρήση στην κλίση του 112. Εκεί να στοχεύει το e-call. Και ε, εγώ έχω μελετήσει και τα δύο συστήματα στο σχέδιο γνωμοδότης. Εάν τελικά στο τέλος της ημέρας καταλήξουμε διαφορετικά, τότε θα έχουμε ήδη διαβουλευτεί και μελετήσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ιδιωτικό σύστημα e-call θα πρέπει να ε, λειτουργεί μόνο με προηγούμενη έγκριση και άδεια του ενδιαφερόμενου και θα πρέπει ο χρήστης να είναι απόλυτα ενήμερος για το έβρος και τη φύση των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο και τις δυνατότητες να σβηστούν από το σύστημα. Ε, πιστεύω ότι θα είναι καλό να μπορέσει να χρησιμοποιεί και το σύστημα 112 όταν του αρνηθεί η πρόσβαση στο ιδιωτικό, στην ιδιωτική πτυχή. Δηλαδή να είναι δεσμευμένα, αλληλένδετα αυτά τα δύο συστήματα. Από το 1995 έχουμε την οδηγία για την προστασία δεδομένων και η οδηγία e-privacy, ιδιωτική, ιδιωτική σφαίρα κλπ. Έχουμε λοιπόν ε, ολόκληρο σύστημα ε, προστασίας δεδομένων το οποίο θα πρέπει να, ε, να μελετηθεί εν μάλιστα μίας αναθεώρησης. Ακόμα υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα εκκρεμή και δυναμικής φύσεως. Καταρχάς ο ορισμός. Τι εννοούμε με ελάχιστο κατόφλι ε, δεδομένων ε, όταν το μεταβιβάσουμε αυτό και το διαθέσουμε στο συστημα ECO. Ποιο είναι το ελάχιστο, το minimum. Επίσης, πώς μπορεί να ληφθεί μία προσωπική έγκριση του χρήστη για τα προσωπικά δεδομένα, για το προσωπικό σύστημα, το ιδιωτικό σύστημα αν θέλετε. Ε, έχουμε επίσης ε, ε, ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε το car sharing, δηλαδή πολλαπλοί επιβάτες, η διαδρομή κλπ υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε για να προστατεύσουμε τα δεδομένα τα οποία θα κυκλοφορούν μέσω αυτού του συστήματος από κλοπή, από hacking και από παράνομη χρήση. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ τις νομικές πτυχές ε, για να ενσωματωθούν μέσα στην ε, γνωμοδότηση αυτή, μέσα στην ιδέα αυτή, μαζί με όλες τις πτυχές της προστασίας δεδομένων. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου τώρα, μιλάω επί της διαδικασίας, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου έχουμε χρόνο για τις τροπολογίες, και στις 18 όπως αρχικά είχα την πρόθεση μπορούμε να ψηφίσουμε στις 18 12 όταν είχαμε ολοκληρώσει την έκθεση, οι συγητές των άλλων πολιτικών ομάδων δεν είχαν οριστεί και η ΙΜΚΟ ήδη στις 6 ήθελε να ψηφίσει. Εμείς είχαμε αντίρρηση διότι θέλαμε να ληφθεί υπόψη και δική μας γνωμοδότηση. Ανέβαλα λοιπόν την ψηφοφορία για τον Φεβρουάριο, οπότε έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και πιστεύω ότι είναι καλύτερο εμείς να καταλήξουμε εδώ για να μπορέσουμε εν συνεχεία να, τη δώσουμε και στην ΙΜΚΟ. Ε, η προστασία των δεδομένων περιορίζεται ε, στο άρθρο 6, ό,τι δηλαδή έχει σχέση ε, με, την, με, νομική, με τα νομικά δεδομένα και με τα, ε, με τα αιτιολογικά 8 και 13 άρθρο 6 και το λογικά 8 και 13. Ε, μπορεί να είναι μικρό το εύρος των νομικών στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό. Σημαντικό. Ε, θα πρέπει λοιπόν εδώ αυτό το σύστημα e-call να συνοδεύεται από από μέσα προστασίας δεδομένων, αλλά δεν θα έχει την ίδια ισχύ και το ίδιο εύρος όπως μια βασική οδηγία προστασίας δεδομένων. Γι' αυτό πιστεύω ότι προτιμώ να βασιστώ στο άρθρο 49 αντί στο άρθρο 50. Αλλά οι άλλοι εισηγητές και η Επιτροπή, αν θέλει, ντε και σώνει το άρθρο 50, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Οπότε εδώ επισέρχονται θεσμικά και πολιτικά ζητήματα. Αλλά απόψε περιεχομένου και ουσίες δεν μου φαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο να κολλήσουμε σε αυτό το θέμα των, άρθρων πιο... Ε, δεν νομίζω να υπάρχουν ε, προ, προσκόμματα και μπορούμε να δώσουμε μια γνωμοδότηση από τη ΛΥΠΕ χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ. Έχουμε διάφορους ομιλητές. Η κυρία Ιντβέλτ, πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή που δούλεψε τόσο γρήγορα, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτό το πρώτο σχέδιο κειμένου. Υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα που θα ήθελα να θίξω. και επί των οποίων έχω κάποιες ανησυχίες. Καταρχάς για θέματα προστασίας δεδομένων. Λέτε ότι δεν θα αποθηκευθούν δεδομένα, δεν θα υπάρξει ανείχνευση των δεδομένων, αλλά με τόσες άλλες πολλές περιπτώσεις είδαμε ποια είναι η τάση. Η τάση είναι να επεκταθεί η χρήση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δεδομένα, κάποιος λέει «Α, ενδιαφέρον, ας τα χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο». Και τέτοια δεδομένα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ας πούμε, για τους ασφαλιστές. Όχι κατά ανάγκη προς όφελος των ασφαλισμένων. Γιατί μπορεί να μην αποθηκευθούν αρχικά οι σένσορες, αλλά μπορεί τεχνικά να είναι δυνατόν να αποθηκευθούν και μετά να δει κάποιος να κάνει ένα προφίλ της συμπεριφοράς κάποιου. Μπορεί να ενδιαφέρει τους ασφαλιστές, ε, διάφορους ε, εμπορικούς φορείς. Ακόμη μπορεί να είναι ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία και για την επιβολή του νόμου. Και δεν νομίζω ότι τα θέματα προστασίας των δεδομένων εδώ είναι ίσονο σημασία. Πρέπει πάντα να κοιτάμε γιατί προτάθηκε κάτι τέτοιο. Για να σώσουμε ζωές. Δεν θέλει κανένα βέβαια να φέρει αντίρρηση σε κάτι τέτοιο, αλλή Αλλά το αν για να σωθεί μια ζωή εξαρτώμεστα από ένα κάρο άλλα πράγματα, δεν σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, ότι γίνεται μια τέτοια κλίση και αμέσως στάνει ένα ε, ασθενοφόρο μέσα σε λίγα λεπτά. Εξαρτάται. Θα είναι διαθέσιμο το ασθενοφόρο κτλ. Θέλω, θέλω να κρατήσουμε τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές για να δούμε αν θα σώσουμε παραπάνω ζωές χάρη σε αυτό. Για τα διαδικαστικά θέματα επίσης θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Και για το άρθρο 49 και το άρθρο 50 νομίζω ότι αξίζει να έχουμε την διαδικασία του άρθρου 50. Οι επιπτώσεις ε, στην ιδιωτική σφαίρα είναι αρκετά σοβαρές και υποθέτω θα υπάρξουν και σε άλλες επιτροπές όλο και περισσότερα θέματα όπου θα υπάρχουν τρομακτικά ζητήματα προστασίας των δεδομένων και επομένως θα χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι η συνέπεια του γεγονότος ότι ζούμε σε έναν κόσμο που χρειάζεται όλο και περισσότερα δεδομένα. Επομένως η διάσταση αυτή των δεδομένων και της προστασίας τους γίνεται όλο και πιο σημαντική. Θα πρέπει ε, κάθε φορά να βρούμε έναν τρόπο να μην παλεύουμε για τη διαδικασία του άρθρου 50 να έχουμε μια διαδικασία όπου εμπλεκόμαστε από την αρχή α, για όλους αυτούς τους φακέλους, για όλα αυτά τα θέματα, όπου μπαίνει η διαδικασία του άρθρου 50. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω στείλει δύο σειρές από ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις. Αν, ας πούμε, έχουμε βάλει στο αυτοκίνητό μας ένα τσιπάκι, είναι ενσωματωμένο, αυτό στέλνει συνέχεια δεδομένα. Μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι η σύνδεση γίνεται μόνο όταν υπάρξει ατύχημα. Πότε διαβιβάζει δηλαδή, δεδομένα το τσιπάκι. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της συνέχειας. Θα λάβει κανείς βοήθεια στο, μετά το ατύχημα αν τη χρειάζεται. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι προετοιμαζόμαστε και ότι δεν θα επιτραπεί η συνεχής παρακολούθηση των οδηγών. Μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα, χρησιμοποιείται από εμπορικούς φορείς για σκοπούς που δεν θέλουμε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι τέτοιο. Οι πράσινοι πιστεύουν ότι η έκθεση του κυρίου Φως πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα θέλαμε να μας δοθούν κάποιες εγγύησεις. Γι' αυτό σκοπεύουμε να υποβάλουμε διάφορες τροπολογίες. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου να μπορεί να σβήνει το e-call, να το κλείνει. Και όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές, όλα τα apps, θα πρέπει για αυτά να προσυπογράφει ο ιδιοκτήτης. Ή όταν, ας πούμε, υπογράφει μια, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο επόπτης προστασίας των δεδομένων μας εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέσα προστασίας για την ιδιωτική σφαίρα των οδηγών. Δεν υπάρχει επαρκή προστασία. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας. Υπάρχει το θέμα της ανείχνευση, της ανείχνευση δεδομένων. Θα πρέπει να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα και αν υπάρχουν επίσης τα δεδομένα, διάφοροι φορείς μπορεί να ενδιαφερθούν να τα χρησιμοποιήσουν, προφανώς. Θα πρέπει να, να προστατεύσουμε τους οδηγούς από κάτι τέτοιο για τους χρήστες του e-call. Και ένα τελευταίο. Δεν πιστεύω ότι ο εισηγητής ε, μπορεί να αποφασίσει αν η άλλη επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το άρθρο 49 ή οποιοδήποτε άλλο άρθρο. Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσουμε, να το συζητήσουμε τώρα αυτό εδώ. Είμαι σκιώδη εισηγητή και συντονίστρια και στη συνάντηση των συντονιστών την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την έκθεση. Οι πράσινοι θεωρούν ότι το άρθρο 50 είναι σημαντικό. Δεν είναι ίσονο σημασία η απόφαση αυτή. Αφορά την προστασία των δεδομένων και την προστασία του ιδιωτικού βίου και της ιδιωτικής σφαίρας τεράστιο θέμα για την Επιτροπή μας. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι παίζουμε το ρόλο μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Ευχαριστώ την κυρία Σαρτζεντίνη. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Φως που το διευθέτησε το θέμα, παρουσίασε το σχέδιο γνωματός τόσο γρήγορα και τόσο καλά. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι εδώ έχουμε δύο ε, πτυχές. Επίγουσες περιπτώσεις, ιδιωτική χρήση. Ε, και επίσης εδώ υπάρχει και το θέμα της ανείχνευσης της ε, τοποθεσίας που βρίσκεται, παρακολούθηση του, της πορείας κλπ. Άρα αυτή, αυτά τα δεδομένα πρέπει πράγματι να μην χρησιμοποιούνται να είναι εν υπνώση. Ε, και να ενεργοποιούνται μόνο σε περίπτωση ε, ανάγκης, απόλυτης ανάγκης. Πρέπει να αποφύγουμε την χρήση για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς στους οποίους στοχεύουμε, διότι θα μπορούσαμε ε, να φανταστούμε μια κατάσταση όπου όλες αυτές, οι υπηρεσίες και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, δεδομένου ότι ε, θα υπάρχει και ένα τέλος, ε, μια συνδρομή, ένα κόστος ε, στη χρήση των υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αξιολόγηση και να μην μπλέξουμε σε δυσάρεστες παρενέργειες. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία αναφέρει στο σχέδιό του είναι πάρα πολύ σωστά, εύλογα και απλώς θα πρέπει να προσέξουμε να αποφύγουμε τις παρενέργειες που ανεπιθύμητες. Είναι επίσης σωστό και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ε, τις δύο αυτές υπηρεσίες ε, έτσι ώστε ο χρήστης ε, να μπορεί διαχειρός να απενεργοποιήσει ε, το e-call, την υπηρεσία αυτή, όποτε επιθυμεί. Αυτή είναι και η θέση μας. Για μας το άρθρο 50 έχει ιδιαίτερη σημασία και μένουμε σε αυτό. Κύριος Κίκοφ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα τον κύριο Φως από την αρχή. Έχω ανησυχίες, πολύ άριθμες ανησυχίες. Θα επικεντρωθώ σε αυτές που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, γιατί πρόκειται μόνο για γνωμοδότηση. Ε, δυστυχώς ε, βρίσκομαι στην ε, περίεργη θέση, ζηλευτή θέση, να συμφωνώ με την κυρία Ιντβέλτ δύο φορές σήμερα δεν υπάρχουν ε, σαφές παράμετροι ή σιγουριά για το, τη χρήση που μπορεί να γίνει σε αυτές τις συσκευέ. Ε, πάντα είμαι κοινικός για αυτά τα θέματα. Ε, για θέματα... Για... Τι γίνεται με τους κομπιούτερς δηλαδή και πώς σταματάς κάποιον ε, από να χρησιμοποιήσει παράνομα ας πούμε κάποια πράγματα και να παραβιάσει τον νόμο. Παραδείγματο χάρη στους ε, γερμανικούς αυτοκινητόδρομους, πώς τους εμποδίζεις ε, τους Γερμανούς να ε, τρέχουν σαν τρελή ας πούμε, που δεν υπάρχει μια και δεν υπάρχει όριο. Έχουμε θαυμάσει ιδέες και χαίρομαι, ε, κύριε Φως, ε, για όλα όσα είπατε, όσα άκουσα. Ε, τον ε, χειρίζεστε με μεγάλη δεξιοτεχνία αυτό το φάκελο, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν τρομακτικά θέματα προστασία των δεδομένων εδώ. Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο, με, η μετριοπαθής χρήση ε, και η προστασία αυτών των δεδομένων. Θα συλλέγονται, ας πούμε, από τους... Ε, δεν θα συλλέγονται από φορείς, αλλά από μια συσκευή, εμπορική συσκευή που πουλιέται μαζί με το αυτοκίνητο. Ε, καταλαβαίνετε τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν. Θα είναι ε, ακριβό, παραγωγικό και διάφορες οργανώσεις ε, εκφράζονται με μεγάλη έμφαση. λένε ότι Τελικά ποιος είναι ο υπεύθυνος, ο κατασκευαστής ας πούμε. Η παραγωγή δεν είναι σωστό να, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε μια συσκευή για οποιοδήποτε έλεγχο. Επίσης, για τη συλλογή των δεδομένων, όπως είπαμε και για άλλα θέματα, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο αναλογικό και εφόσον είναι αναγκαίο. Αυτή η πρόταση πιστεύω ότι είναι περιττή και η συλλογή δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο είναι εντελώς περιττή παραβίαση και δίζηση στην ιδιωτική σφαίρα των ανθρώπων. Ο κύριος Ντεϊόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ελέγχθησαν, πάρα πολλά, τα οποία με βρίσκουν και ε, σύμφωνο εμπολής. Παρακολουθώ πολύ καιρό αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και όταν σταθήκαμε στα τεχνικά στοιχεία, η κυρία Ιντβέλτ ε, τόνισε τη σκοπιμότητα του ζητήματος λέγοντας ότι υπάρχουν ορισμένες ε, ουσιώδεις δυσκολίες. Η μόνη χώρα που είχε κάποια εμπειρία επί του θέματος ήταν η τσεχική δημοκρατία και είχε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την λήψη των σημάτων, του σήματος. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά ξέρω ότι χρειάζονται άλλες τεχνικές προδιαγραφές και αλλαγές, έτσι ώστε ε, να μπορέσουν τα νοσοκομιακά να βρεθούν ακριβώς στον τόπο του ατυχήματος. Το σύστημα θα πρέπει να έχει ενιαίο χαρακτήρα στην Ευρώπη δηλαδή να υπάρχει ενιαία εφαρμογή και νομίζω ότι από τεχνικής πλευράς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Νομίζω ότι υπάρχουν μείζωνα προβλήματα σε σχέση με τη λήψη του σήματος και πολλοί πολίτες ανησυχούν και μας λένε «Μα στο όχημά μου ε, έχουν εγκαταστήσει ένα μέσο να τσιπάκι το οποίο μπορεί να με παρακολουθεί και πατού, να με κατασκοπεύει επί της ουσίας. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους πολίτες. Δεν θα πρέπει να δίνουμε την εντύπωση σε αυτή τη γνωμοδότηση ότι εκτός από το 112 υπάρχουν και άλλες ε, δυνατότητες για αντιμετώπιση μιας επίγουσας ανάγκης. Δηλαδή, η χρήση δεν είναι ίδια με την κλίση του 112. Υπάρχουν πολλοί φόβοι και ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από τους πολίτες. Ο μεγάλος αδελφός είναι πανταχού παρόν, αυτό μας λένε. Και αναρωτιόνται κατά πόσο θα ε, περιοριστούμε στον εντοπισμό και μόνο. Θα πρέπει να ξέρουμε επακριβώς τι συμβαίνει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι πολίτες ε, ανησυχούν και εκφράζουν τους φόβους τους και εμείς ήμασταν ε, αρκετά επικριτικοί ως ομάδα. Εάν ε, υπάρχει επίγουσα ανάγκη, καλούμε το 112. Το σύστημα αυτό έχει βέβαια διαφορετικό στόχο. Μπορούμε να τον συζητήσουμε, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους όπως λέει και ο κύριος ε, Βος στην ε, γνωμοδότηση του, θα πρέπει ο οδηγός να αποφασίσει σαφώς εάν πραγματικά επιθυμεί την ύπαρξη αυτού του σήματος, εάν θέλει να γίνεται η εκπομπή αυτού του σήματος, ναι ή όχι. Επίσης, θα πρέπει να συγκρίνουμε την κατάσταση με τον κανονισμό ε, περί ζωής και, εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχουν ζητήματα αρχής, δηλαδή δεν θα πρέπει να πρόκειται για αυτοματισμούς. Είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζουν θετικά οι πολίτες. Θα ήθελα ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ή εκπρόσωπος των Ευρωπαίων Δημοκρατών να λάβει το λόγο, νομίζω. Του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, με συγχωρείτε, ή εκπρόσωπος. Υπάρχουν ε, μεγάλες ανησυχίες σε σχέση με την ύπαρξη του συστήματος της κλίσης 112 και το πρόβλημά μας είναι ότι πρόκειται για έναν εξοπλισμό όλων των νέων οχημάτων ε, όπου ε, ο μηχανισμός είναι αρκετά παρεμβατικός διότι υπάρχει σήμα εντοπισμού και οι ρήτρε διασφάλισης σχετίζονται με ένα συσχετισμό ως προς το 112. Ανοίγουμε ε, νομίζω το δρόμο σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και πιο διευρυμένες υπηρεσίες, δηλαδή όλες ε, τις υπηρεσίες που έχετε και στο κινητό σας με τον γεωεντοπισμό. Οι υπηρεσίες αυτές, η υπηρεσία αυτή ήδη υπάρχει και η κυρία Σαρτζεντίνη είπε ότι ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο εντοπισμός θα χρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς σκοπούς. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Ήδη έχει ε, προωθηθεί από τους κατασκευαστές ε, ε, οχημάτων ή από, τις διάφορες, από τα διάφορα applications. Άρα αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ίσως ορισμένοι καταναλωτές το επιθυμούν. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να καταπατά την νομοθεσία προστασίας δεδομένων, αλλά θα πρέπει να συμμορφούνται απόλυτα με πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας που σχετίζονται με την κλίση 112 και δεν θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ανείχνευση. Και επίσης το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να συνενέσει σε σχέση με το e-call και την προσθέμενη αυτή αξία. Άρα η ουσία είναι ότι δεν θα υπάρχει γεωεντοπισμός εάν το φυσικό πρόσωπο δεν συνενεί. Θέλουμε δηλαδή να ε, συνενεί το ε, φυσικό πρόσωπο αν γίνει χρήση γεωεντοπισμού. Άρα θα μπορούσαμε είτε να προσθέσουμε κάτι στο άρθρο 6 όπου υπάρχει μια διασφάλιση ως προς την εξίσωση του μηχανισμού με την κλίση 112 ή να υπάρχει ιδιωτικό σύστημα e-call με προστιθέμενη αξία ή θα μπορούσαν οι κατασκευαστές οχημάτων να δεχτούν αυτές τις εφαρμογές, να τις επιτρέψουν και βεβαίως να υπάρξει προστασία προσωπικών δεδομένων όπως ζητά η ΛΥΜΠΕ, διότι δεν θέλουμε να υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την παρακολούθηση των πολιτών. Δεν ξέρω κατά πόσο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ή εκπρόσωπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τον εισηγητή κύριο Βος για το σχέδιο γνωμοδότησης. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες για την ιδιωτικότητα και την ε, νομική ασφάλεια, την νομική προστασία που να συνάδουν με όλο το νομικό πλαίσιο των οδηγιών για την προστασία δεδομένων 95-46 και αυτό ε, περιλαμβάνεται, αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του κειμένου. Όσον αφορά τώρα την προστιθέμενη αξία, η Κομισιόν ε, πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μία εντολή βάσει του όλου πλαισίου για το 112, για τον αριθμό 112 και η Κομισιόν πιστεύει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί αν θέλουμε να ρυθμίσουμε και ιδιωτική χρήση ε, ή άλλους σκοπούς, διότι σαφώς εμπλέκονται σοβαρά ζητήματα προστασίας δεδομένων. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την δυνατότητα απενεργοποίησης του e-call από το χρήστη, η Κομισιόν πιστεύει ότι αυτό θα μπορέσει να περιορίσει σοβαρά, να υπονομεύσει δηλαδή τα ωφέλη ε, για τον ιδιώτη χρήστη του όλου συστήματος. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η βασική επιφύλαξη που εκφράστηκε εδώ, δηλαδή η συνεχής ανείχνευση παρακολούθηση του ηχήματος αποκλείεται ρητός από την αρχική πρόταση της Κομισιόν, το, η οποία απέβλεπε, όπως σας είπα, στην χρήση του e-call για τον αριθμό 112. Όσον σε ό,τι αφορά τώρα το διαχωρισμό μεταξύ του, του, και άλλων χρήσεων που ενδεχομένως να προσφέρουν τη θέμενη αξία, υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες, αναμφίβολα, αλλά το θέμα είναι θα μπορούσαν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν τα ίδια στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε παράλληλη χρήση. Θα υπάρχει δηλαδή μία επικάλυψη χρήσεων την οποία δεν ε, θέλουμε. Ευχαριστώ. Ο Άξελ παρακαλώ, ο εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι το οποίο η Κομισιόν μόλις ανέφερε. Ε, κατ' ουσίαν, ε, όπως προέκυψε και με τη συζήτηση ε, με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ και με την εισηγήτρια του ΙΜΚΟ, ότι θέλουμε να περιορίσουμε το, τη λειτουργία του συστήματος στο e-call 112. 1, 1, 2. Γι' αυτό εγώ ε, ως ε, προκαταβάλλοντας ε, την συζήτηση έχω συμπεριλάβει και την άλλη πτυχή, την ιδιωτική χρήση, διότι πολλές φορές αναφέρεται και θα ήθελα, για να είμαι πολύ προσεκτικός, να το αναφέρω. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το θέμα αυτό στο ΙΜΚΟ μου έχουν διαβεβαιώσει ότι πρόκειται μόνο η call τον αριθμό 112 και τη χρήση του 112. Άρα θα πρέπει να θέσουμε ένα όριο στην χρήση της προστασίας των δεδομένων, μια χρήση, στην μια οροφή στα δεδομένα, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να αποφασίσει εάν το θέλει ή όχι. Γι' αυτό έβαλα και τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Εμείς εδώ δεν στοχεύουμε στην μεταβίβαση ιδιωτικών στοιχείων, απλώς στην διαγραφή ε, δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν χρειάζονται και την απενεργοποίηση του συστήματος. Πιστεύω ότι αυτό είναι, αυτή η δυνατότητα, αν δοθεί, προσφέρει μια καλύτερη χρήση ε, στα δεδομένα. Μόνο σε επίγουσα ανάγκη και μόνο όταν έχει ο χρήστης ενεργοποιήσει το σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το e-call. Αυτή πιστεύω είναι η ουσία του συστήματος και η όλη ιδέα ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η εκπρόσωπος δηλαδή, ε, εξέφρασε την άποψη του φορέα. Και όσον αφορά τώρα το ιδιωτικό σύστημα, την ιδιωτική χρήση, μπορούμε να εκφράσουμε τις ιδέες μας για το πώς θα θέλαμε να διαμορφωθεί στο μέλλον. Ενδεχομένω όμως τώρα αυτό να μην παίξει κανένα ρόλο, να μην, ε, να μην έχει καμία σχέση με το στόχο μας σήμερα που είναι ορισμός 112. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να εν είδη προετοιμασίας ε, και, νομι... επεξεργασίας του νομικού πλαισίου να τα σκεφτούμε όλα αυτά για το μέλλον. Αλλά ακόμα και αν θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτό το, την ιδιωτική χρήση, τότε θα πρέπει ο πολίτης να έχει την ευθύνη να αποφασίσει αν θέλει να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό ή όχι, αν μπορεί να το ενεργοποιήσει ή όχι και εν συνεχεία ο ίδιος έχοντας υπόψη το κόστος, την ασφάλιση, το κόστος χρήσης, το ασφαλιστικό κόστος κλπ. να μπορέσει να εκμετελευσεί μία καλή τιμή, μία ε, σωστή τιμολόγηση του όλου συστήματος. Βεβαίως, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει, θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί μια ενημέρωση, να μπορεί να ξέρει τι είναι το σύστημα, πώς να το χρησιμοποιεί και τι είδους δεδομένα θα κυκλοφορούν ε, όπως προβλέπονται από τις οδηγίες και το πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Όσον αφορά Τώρα, την χρήση, την νομική βάση του άρθρου 49 50 δεν έχω ιδιαίτερο πάθος για το ποιο ε, άρθρο θα χρησιμοποιήσουμε. Εάν περιορίσουμε το όλο θέμα στο 112, τότε μπορούμε να πούμε προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ ότι εμένουμε στο άρθρο 50. Ωραία, ωραία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 50. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς ε, πιστεύω ότι ε, η μελέτη του όλου θέματος ε, δεν, είναι, δεν συνάδει ακριβώς με την περιορισμένη ισχύ του άρθρου 50, αλλά αν ε, ανεμένων δεν έχω, είμαι αρκετά ευέλικτος και ε, μπορούμε να προχωρήσουμε πιστεύω γρήγορα στην πρόθεση του θέματος όσον αφορά την ε, εμπορική χρήση τη ε, χρήση για συναλλαγές, για άλλες χρήσεις εκτός του 112, θα αφήσουμε αυτά στην ΙΜΚΟ. Αλλά και σε αυτό τον τομέα ο κάθε χρήστης πρέπει να έχει συγκεκριμένε ευθύνε. Άρα πρέπει να είναι σε θέση να είναι πλήρως ενημερωμένος για τα δεδομένα και επίσης να μπορεί να το απενεργοποιήσει και απενεργοποιήσει. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Φως. Τώρα, <clears throat> το σημείο αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ε, πρωινή μας ε, συνεδρίαση. Επομένως, θα κλείσω τώρα τη συνεδρίαση και θα ξαναρχίσουμε στις 2 η ώρα το απόγευμα με την κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Εκόνα. Και συνεχεία στις 3.30 θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας μόνοι μας, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αυτό, που αυτό το θέμα που μόλις συζητήσαμε ήταν πάρα πολύ σημαντικό και προβλέπεται η κατάθεση τροπολογιών μέχρι την 5η Δεκεμβρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και θα τα ξαναπούμε στις 2 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ.